Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε. bernd lange sagt der gualtieri soll sich hinsetzen. setz dich hin! πείτε στον Γκουαλτιέρη να καθίσει. Du auch. Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι και εσύ και εσύ. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Η διάσκεψη των Προέδρων σήμερα το πρωί έλαβε μια απόφαση για την απονομή του βραβείου Ζαχάρο για το έτος 2015. Σας ανακοινώνω ότι η διάσκεψη των Προέδρων φέτος θα απονείμει το βραβείο Ζαχάροφ στο blogger Ραΐφ Μπαντάουι από τη Σαουδική Αραβία. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη αυτής της απόφασης. Σήμερα, λόγω της ιδιάζουσης περίπτωσης του κυρίου Μπαντάουι, πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ θαραλέος, εξαιρετικά υποδειγματικός άνδρας που αντιμετωπίζει μία από τις πιο ιδεχθείς πινές που επιβάλλονται στη χώρα αυτή και αντικειμενικά μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει μόνο ως ε, ομό βασανιστήριο. Καλό να απονείμει χάρη ο βασιλέας αμελητή τον κύριο Μπαντάουι να το επιτρέψει να ταξιδέψει για να μπορέσει να έρθει να παραλάβει το βραβείο του. Οι σχέσει μεταξύ των κρατών μελών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωση και των θεσμικών οργάνων της Ένωση με τις χώρες ετέρους εξαρτώνται στην ποιότητά τους και από το πώς τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα οι εταίροι μας. Στην περίπτωση του κυρίου οι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όχι απλώς ε, δεν τηρούνται, αλλά παραβιάζονται κατάφορα και καταπατώνται. Γι' αυτό καλό το βασιλέα της Σαουδικής Αραβίας σήμερα να του απονημιχάρει, να τον αφήσει ελεύθερο, να μπορέσει να επιστρέψει στη σύζυγό του και να έρθει το Δεκέμβριο στο Στρασβούργο για να παραλάβει το βραβείο του. Σας ευχαριστώ πολύ. So, ähm, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Ζήτησε το λόγο η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Uh, uh, Εχθές έθεσα το θέμα του, της φαντασιακής ψηφοφορίας της κυρίας Λεπέν, συμπροέδρου της ομάδας της. Και θα ήθελα να σας πληροφορήσω για τα αποτελέσματα της ερεύνης. Ευχαριστώ την υπηρεσία της Ολομελίας για την επαγγελματικότητά της και τη γρήγορη αντίδρασή της και θα ήθελα να ζητήσω από τον Πρόεδρο να χρησιμοποιήσει πλήρως το άρθρο 176 και 177 του κανονισμού που λέει ρητά ότι η ψηφοφορία είναι αυστηρά προσωπική και ότι ο κάθε βουλευτής 166 και 167 και ότι ο κάθε βουλευτής είναι υπεύθυνος για την ψήφο του. πλασματικής μάλλον ψηφοφορίας. 166 και 177. Κύριε Λεπέν, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, τη απουσία μου εχθές με κατηγόρησαν τελείως άδικα ο κύριος Βέμπερ με κατηγόρησαν για πράξεις που δεν διέπραξα και αυτό αποκαλύφθηκε στη διάσκεψη των Προέδρων σήμερα το πρωί. Ο κύριος Βέμπερ διέπραξε δύο αδικήματα και τα δύο ψευδή δηλώσεις, χωρίς καμία απόδειξη, δυσφήμιση. Τι έγινε λοιπόν εχθές που εξηγεί αυτά τα, αυτούς τους θεατρινισμούς. Βγήκα αφήνοντας την κάρτα μου όπως κάνουν δεκάδες βουλευτών που την ξαναπαίρνουν στο τέλος της συνεδρίασης. Ε, ακούστε, αυτά είναι τα μόνα που έχετε να πείτε. Α, ο συνάδελφος Δεκράμπ που είναι τελείως άμεμπτος και άψογος θεώρησε ότι έφυγα για λίγα λεπτά και έκανε τέσσερις ψηφοφορίες στη απουσία μου, τέσσερις. Και, και χωρίς να μου ζητήσει την άδεια. Και χωρίς να μου ζητήσει την άδεια. Επαναλαμβάνω, και χωρίς να μου ζητήσει την άδεια. Πράγματι αυτό ήταν, δεν ήταν άψογο. Αλλά αυτό δικαιολογεί, δικαιολογεί λέγω, αυτά που κάνατε, κύριοι συνάδελφοι. Θεωρώντας ότι θα επέστρεφα σε λίγο, επέδειξε και πνεύμα υποσύνης, υποτικότητος. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, θα δω τι θα κάνω και θα καταθέσω μήνυση κατά του κυρίου Βέμπερ, ο οποίος εξέφρασε απαράδεκτες κατηγορίες για μένα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα απασχόλησε το θέμα αυτό τη διάσκεψη των Προέδρων. Ο κύριος Βέμπερ έχει το λόγο επί προσωπικού. Κύριε Πρόεδρε, Μιλήσατε κυρία ο κύριος Βέμπερ τώρα. Ακούγοντας αυτές τις δηλώσεις έχουμε μείνει άναυδοι. Είναι το απάβγασμα του θράσους και της ανέδειας αυτά που ακούμε σήμερα εδώ μέσα. Κυρία Λεπέν, γνωρίζουμε ότι εσείς δεν ξέρετε, δεν σκαμπάζετε από κανονικές δημοκρατικές διαδικασίες. Τα ξέρουμε όλοι εδώ μέσα αυτό. Να σας κάνουμε κάνα φροντιστήριο. Στη δημοκρατία την εντολή που λαμβάνουμε από τους πολίτες, εμείς τη θεωρούμε ιερή. Είναι ιερή εντολή. Και όταν έχεις μια ιερή εντολή, αυτή η εντολή, δημοκρατία σημαίνει να ακούς και τον άλλον, κυρία συνάδελφε, Λοιπόν, στη δημοκρατία λέγω είναι ιερή εντολή μας, την έχουν αναθέσει οι πολίτες, οι ψηφοφόροι. Και αυτή η εντολή δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται σε κανέναν άλλον σε κάποια κράτη-μέλη αυτό είναι αξιόπινη πράξη. Είναι κακούργημα και μπορεί κανείς να προσφύγει στο δικαστήριο. Ευτυχώς για εσά, στην Ευρώπη αυτό δεν ισχύει σήμερα. εμεί το θεωρούμε ιερό αυτό το καθήκον της εντολής. Εδώ έχετε ένα μεγάλο σκάνδαλο στις πλάτες σας και υποστηρίζουμε τον Πρόεδρο και τον καλούμε να λάβει κάθε ε, νόμιμη δράση εναντίον σας. Meine Damen und Herren, heute Morgen war... Κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωί το συζήτησε το θέμα αυτό η διάσκεψη των Προέδρων και ε, θα γίνει η αντίστοιχη εξέταση στο Προεδρείο που είναι το αρμόδιο όργανο. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ μπορεί να είναι βέβαια ότι θα λάβουμε υπόψη όλα τα σχετικά άρθρα του κανονισμού. Έχουν διανεμηθεί τα χτεσινά πρακτικά, τα συνοπτικά. Διαφωνεί κανεί με τα κείμενα.